I'm trying to start. Colleagues, can, can we start now? Because can we start? Can we start, please? Because I know that members. Μπορούμε να ξεκινήσουμε παρακαλώ γιατί γνωρίζω πως ορισμένοι συνάδελφοι έχουν και άλλες ε, υποχρεώσεις. Δώσω το λόγο στην ε, συνάδελφο Βερνάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, πρόκειψαν κάποιες αλλαγές, ειδικά σε ό,τι φορά το άρθρο 14 για τον τρόπο παρουσίασης. Συμφωνήσαμε με το ΕΛΚ για να έχουμε ένα μέγεθος ε, ελάχιστο ανάλογα με το μέγεθος της συσκευασία 1,2 mm έω 2,5 μιλιλέτρου για πάνω από 75 σαντιμέτρου τετραγωνικά εκατοστά τώρα για το θέμα της ε, παρουσίασης ε, και δεν μπορούσαμε να βρούμε συμφωνία που ικανοποιεί όλους, ο καθένας μας έχει κάποιες αρχές ε, και ορισμένες φορές δεν μπορούμε να τις παραβούμε. Υπήρξε λοιπόν συμβασμό με το ΕΛΚ για την παρουσίαση με γραφική μορφή εναρμονισμένη μέσω επιτροπολογία σε όλες τις ευρωπαϊκέ χώρες με τη δυνατότητα για ορισμένα κράτη να διατηρήσουν επιπλέον τα εθνικά σχέδια εάν δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Αλλά δεν συμφωνήσαμε σχετικά με τις ε, βασικές προφορίες ενέργεια, λύπη, γλυκίδια, ε, ζάχαρη κλπ. να αναφέρονται στο εμπρόσθετο τομέα του συσκευασίας τώρα σχετικά με το 29 ένταξη ενέργειας λοιπόν ε, ε άλατος ε, κορεσμένο λύπη ίνες και πρώτε πρωτεΐνες αυτές οι αναφορές είναι υποχρεωτικές. Δεν συμφωνήσαμε λοιπόν όμως με το σημείο στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται αυτές οι ενδείξεις. Αλλά είπαμε πως θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνονται στο ίδιο σημείο. Έχουμε εννέα συμβαστικές ε, ε, συμβαστικές λύσεις με το ΕΛΚ και το ΑΛΔΕΚ κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουν τα βασικά σημεία του κειμένου, καλύπτοντας ε, μια σειρά τροπολογιών που ζητούσαν τη διαγραφή κάποιων σημείων που είχε καταθέσει ο κύριος Καράς σχετικά με το γράφο της Επιτροπής τώρα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτών των ψηφοφοριών θα μπορεί να είναι ισόρροπο, θα διασφαλίζει καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνουν υπόψη κάποια σημεία που είναι προβληματικά για τους παραγωγικούς, εξαιρέσεις για τα αλκοολούχα ποτά και για τα μη προσυσκευασμένα. Αυτά. Τώρα, οι συμβαστικέ τροπολογίε που είχαμε, στο πίσω είχαμε καταλήξει την περσμένη εβδομάδα, συμφωνήσαμε με το άρθρο 8 τη ε, θέμα των ευθυνών δεν υπήρχε ουσιαστικό πρόβλημα εδώ, αλλά καταψηφίσαμε όλες τις τροπολογίες καράς. Για το άρθρο 9, υποχρεωτικέ προφορίες, φυσικά πήραμε την ε, πρόταση της Κριστέλ για την ημερομηνία κατασκευής και την ενδεχόμενο κατάργηση της λίστας με τις επιτροπολογίες για το άρθρο 20. Αξαιρέσαμε τα αλκοολούχα για μια τριετή περίοδο και για πενταετή περίοδο συμπεριλαμβανομένου και το ίνου και των ίνων των ματιδών φωτών βρήκαμε την ε, και θα πρέπει να αναφέρεται η έκφραση ανά 100 γραμμάρια σε όλες τις ε, συσκευασίε. Για τα μη προσκευασμένα προϊόντα παραμένει το, τα ε, αλλεργιογόνες ουσίες, συνθήκες αποθήκευσης, χώρα καταγωγής, αλλά οι τρόποι ανακοίνωση τη προφόρησης έγιναν πιο ευέλικτες. Μιλάω για τα μη προσκευασμένα, ε, επί μια ετικέτας, σύμφωνα με τις εθνικέ διατάξεις που θα ανακοινωθούν στην Κομισιόν. Κατά τα υπόλοιπα δεν είχαμε προβλήματα, διότι οι τροπολογίες του κ. Στεναρής γίνανε αποδεκτές, ο κ. Σνεμπή δεν κατά τις τροπολογίες και άρα δεν προέκυψαν προβλήματα. Συνολικά λοιπόν νομίζω ότι όλοι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε στην περαιτέρω ενημέρωση του καταναλωτή. Ευχαριστώ. Uh, Εντάχει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ο Χίτον Χάρης είναι στην Αμερική αυτή τη βδομάδα αλλά είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Βεγνό και υποστηρίζουμε όλες τις ε, τροπολογίες συμβασμού. Ωραία. Ωραία, θα είναι απλή η διαδικασία. Ας ε, συνεχίσουμε. Άρθρο 1, 48, Κάρας, ποιοι είναι υπέρ. Η κυρία Βερνιό. Μία μόνο διευκρινιστή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βοηθούς και την ε, γραμματεία που μας βοήθησαν στις τροπολογίες που δεν ήταν ε, ιδιαίτερα εύκολες. Ωραία. Θα προσπαθήσω να μην προχωρώ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 48 κάρας. Δι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 κάρας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ηλεκτρονική ψηφοφορία σας παρακαλώ. Υπέρ. Α, όχι, λέει. Εφόσον γίνεται ηλεκτρονική. Έχετε όλοι οι κάρτες. Έχετε όλοι οι ηλεκτρονικές κάρτες. Έχετε όλοι κάρτες. Λοιπόν, θα κλείσω την ψηφοφορία. Πέρας. 23 υπέρ, 18 κατά, ένας, μία αποχή άρα εγκρίνεται. Ορισμοί 51 κάρα υπέρ. Α, θα είναι διαφορετική η πλειοψηφία. Κάρτες και πάλι. Να δω τι μεταλλάξεις γίνονται. 16-26. Απορρίπτεται. 52 κάρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές επίσης απορρίπτεται 55 δεν ψηφίζουμε την 55 56 57 μαζί υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές επίσης απορρίπτεται σαφώς 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 4 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άρα ψηφίζουμε την 71-72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 73. Όχι, λέει πρόεδρος. 73, 70, Η 70 απορρίφθηκε. No, we didn't need to do 72? No, we don't. Μα τι ψηφίσαμε την 72. Υπέρ. Ναι, αυτό είπα και εγώ, ότι 70 απορρίφθηκε. Έχω δύο συμβούλου αυτή τη στιγμή. Τώρα τι ψηφίζουμε, λέει η πρόεδρος. Α, την 72, υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα πάμε στο συμβασμό 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 10. 90 και 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 91 υπέρ. Κατά. Ξανά σας παρακαλώ. 89-90 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 91 κάρας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα τώρα πάμε, επειδή εγκρίνεται πάμε στις 95-96 τον χάρη του Μπον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία συμβασμού 3 υπέρ κατά αποχές ε, σαφώς εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 107. Άρθρο 16, τροπολογία 107. Υπέρ της 107, δι, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται, 108, χιτον χάρις υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρθρο 17 110 κάρας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται βερνιό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 κάρας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 κάρας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού 4 υπέρ κατά αποχές σαφώς εγκρίνεται. Άρα πάμε στην 120. Άρθρο 21. Κάρας 120 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επίσης άρθρο 22, 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 23 κάρας 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 25 126 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 29 συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σαφώς άρα φτάμε, φτάνουμε στο, στην 127 λέει α όχι όχι με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος κα. 152 διορθώνει η πρόεδρος άρθρο 30 τροπολογία 152 Κάρας Α, ο, ο κύριος Κάρης ήταν πολύ απασχολημένος. Υπέρ της 152. Υπέρ, είπα. Κατά. Απορρίπτεται. 153. σαλτεμός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 μετά πάμε. 19. Βερνιό υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 155 σαλντεμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 εκπίπτει. Άρα πάμε τώρα στο 20, την 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα πάμε στο άρθρο 33 Τροπολογία Κάρας, 163 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 34, 165 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 22 βερνιό υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 164 σβάμπ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 166. Σαλδεμός υπέρ. Υπέρ, υπέρ σας παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Γιατί δεν ψηφίζετε ως ομάδες. Λοιπόν, 166. Σαλδεμός Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. 21. Α, απορρίπτεται. Ισοψηφία. 21-21. Sorry, sorry, I couldn't help you with that. 167. Χίτον Χάρις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Yes, they were all rejected, that's right. Okay, 168. 168. Χίτον Χάρις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Όχι, δεν το έχω αυτό το σημείο στη λίστα μου. Άρα το πρώτο τμήμα αφορά τις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Άρα εγκρίθηκε ολόκληρη η τροπολογία. Φτάνουμε στον συμβασμό 8, στο άρθρο 35, υπέρ του 8. Κατά αποχές εγκρίνεται σαφώς. Άρα οι άλλες καταπίπτουν 174. 174 μαζί με την 175 και 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Βερνιό 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 174, 175, 179 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 181 χίτων χάρη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 184 και 175 μαζί υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτονται. Να ελέγξω ή να μην ελέγξω, λέει η πρόεδρο. Ωραία, σε ελέγξουμε. Νομίζω ήταν σαφέ, αλλά μερικοί δεν ψήφισαν. 174 και 175. 174 και 175. Απορρίφθηκαν σαφώς. 182 Σαλτεμόζ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 183 Χίτων Χάρης υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 184 Κάρας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 185 και 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 185-186 στο άρθρο 38 όμως αυτή τη φορά υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 187 καταπίπτει τότε. Άρθρο 39, 185-186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 40, 185-186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Άρα πάμε στον συμβιβασμό 9, στο άρθρο 41, υπέρ παρακαλώ του συμβιβασμού, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 40, άρθρα 42 και 43 υπέρ, λέει η Πρόεδρος, κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρα 44 έω έως 47, 195-196 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 53, 197, 197 μόνο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 198 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παραρτήματα 199 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 200 Βάις Γκέρμπερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 199 Κάρας υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 199 τμήμα 3 ως προσθήκη ως προσθήκη υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 202 Γκέρμπερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα 199 τμήμα 4 ως προσθήκη κάρας υπέρ, κατά αποχές σαφώς απορρίπτεται. Παράρτημα 2. Ψηφίζουμε όλες τις ε, τροπολογίες Χίτων Χάρης υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 206 κάρας υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται παράρτημα 3 κάρας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 κάρας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 βερνιό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 σαλδεμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράρτημα 4. Ξεχωριστή ψηφοφορία για την 10, τμήμα 1. Χωρίς να αναφέρουμε το chewing gum, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για τις τσίχλες, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται η 10, παράρτημα 5 τώρα. Παράρτημα 5. 220. κάρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 221. κάρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30. Βερνιό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράρτημα 6. Κάρας 222 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31. Βερνιό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά θα το δούμε ηλεκτρονικά ελέγχουμε 224 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 17-26. Πολλές φορές δεν σηκώνετε τα χέρια σας, γι' αυτό είναι δύσκολο να γίνει καταμέτρηση. Λοιπόν, απορρίπτεται σαφώς. 225. Κάρας, υπέρ. Κατά. Α, απορρίπτεται, λέει η Πρόεδρος. 226 και 227 μαζί, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 228 κάρας, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 Βερνιό υπέρ κατά επίσης ελέγχουμε ηλεκτρονικά γιατί είναι ξεχωριστή αρχίζει η ψηφοφορία για την 32 20 υπέρ 22 κατά, άρα απορρίπτεται. Παράρτημα 11. 229 υπέρ. Κατά αποχές 229. Να ελέγξουμε. 229. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται 21 έναντι 19. 230 κάρας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231-232 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Παράρτημα 12. 233 και 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Παράρτημα 13. 236 και 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 235 τμήμα 2 κάρας υπέρ κατά Αποχές ε, απορρίπτεται. 237 κάρας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 238 εκπίπτει, άρα πάμε στο προήμιο. 33 χίτων χάρης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 βενιό υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε, θα την ελέγξουμε και αυτήν ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 1 Βερνιό 20 υπέρ 23 κατά. Άρα απορρίπτεται και τον Χάρης 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 35 χίτων χάρις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 έγινε αποδεκτή, άρα δεν βλέπουμε. 41 ε, μπέρκ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά θα την ελέγξω την 44. Ελέγχουμε την 44. Πέρας. 23 υπέρ, 20 κατά. Άρα εγκρίνεται. 45 σαλδεμός υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά αποχές επίσης εγκρίνεται τελική ψηφοφορία τώρα να γίνει ηλεκτρονικά καλύτερα αρχίζει η ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσατε όλοι ωραία εγκρίνεται ομόφωνα 43 υπέρ κανένας κατά καμία αποχή θαυμάσια κυρία Βερνιό συγχαρητήρια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 Θα ψηφίσουμε την έκθεση Μος. Η συγγήτρια θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες μας ε, επί της ε, έκθεσης ε, των περί τυχερών παιχνιδιών είχα πει πως θα ήταν δύσκολο να εξευρεθούν ορθές λύσεις ε, και αυτό πράγμα αποτοπίθηκε διότι οι θέσεις δίσταντο σημαντικά αλλά είμαι τελικά ευτυχής που είχα τη δυνατότητα να συζητήσω αυτό το σημαντικό ζήτημα με τους συναδέρφους ε, και όχι μόνο διότι είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί αυτή η αγορά προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικότερα οι καταναλωτές και αν ε, τελικά οι έχουν αίσιο πέρας θα έχουμε οδηγηθεί σε, μια πολύ, σε ένα πολύ ισόρροπο αποτέλεσμα και η συνεργασία πραγματικά μερικές φορές ήταν επίπονη ο κύριος Χάρμπουρ να ευχαριστήσω την Κριστέλ Σόλμος για τις ε, συζητήσεις που είχαμε αλλά όπως είπε και η ίδια ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε συμφωνία Βρίσκω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα σε ό,τι αφορά τα μέλη της ε, ομάδας μου αποφασίσαμε ότι το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε, να συντάξουμε και μια έκθεση της μειοψηφίας, κάτι το οποίο θα υπογράψουν ε, διάφοροι στάλφοι και τουλάχιστον ένα μέλος από την ομάδα ALDE. Θεωρούμε πως αυτή η έκθεση δεν, είναι, δεν επιφέρει την κατάλληλη ισορροπία, διότι Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το πεδίο το οποίο μας είχε απασχολήσει από την αρχή. Οι αρχές της ε, ενιαίας αγοράς δεν τηρούνται απόλυτα σε κάποιες τροπολογίες. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις ε, που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η γνώμη της ε, μειοψηφίας. Θα υπάρξουν δύο Κατάλογοι ψηφοφοριών. Ο ένας θα στηρίζει την άποψη αυτής της μειοψηφίας και ο άλλος ε, κατάλογος την έκθεση της κυρίας ε, εισηγήτριας και θα προτείνουμε ένα διαφορετικό ένα εναλλακτικό κείμενο στην Ολομέλεια. Πάντως ε, συμφωνούμε με τα περισσότερα από τα όσα είπε και έπραξε η κυρία Σόλτερ Ευχαριστώ. Διάφοροι συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Παρακαλώ, ας μην ξεκινήσει τώρα συζήτηση, κυρία Γκέπαρτ. Ναι, Όχι, δεν πρόκειται να προχωρήσω σε συζήτηση επί της ουσίας. Αυτή έγινε χθε. Η πολιτική μου ομάδα έχει μία ενιαία θέση και αυτό είναι θετικό. Εμείς δηλαδή υποστηρίζουμε απολύτως το έργο της εισηγήτριας. Βεβαίως σέβομαι το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις Ωστόσο δεν μπορώ να δεχθώ μία εντό εισαγωγικών μομφή. Δεν πρόκειται καθόλου για έκθεση που στερείται ισορροπίας. Είναι εξαιρετικά ισορροπημένη και ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια διότι κατόρθωσε να συμπεριλάβει απόψεις από πολύ διαφορετικές πολιτικές ομάδες όπως των, ε, της, Ηνωμένης, της Ηνωμένης Αριστεράς, των Πρασίνων, της Σοσιαλιστικής Ομάδας και ορισμένων εκ του Λαϊκού Κόμματος και πραγματικά υποκλίνομαι στην ικανότητά της. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θα λάμβανα το λόγο αν δεν άνοιγε, άνοιγε η συζήτηση. Θα ήθελα να πω ότι δέχομαι τη θέση της σκιώδους της κυρίας Κορχόλα και θεωρώ ότι εάν ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή θα έχουμε μία εξισορροπημένη θέση. Εμείς οι Πορτογάλοι έχουμε σαφείς ιδέες ως προς τα τυχερά παιχνίδια και προσεγγίζουμε τη γαλλική θέση. Δεν δεχόμαστε λοιπόν να να δημιουργηθούν παράλληλες πολιτικές ενδοκινοτικά δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μια κοινωνική πολιτική, όπως ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ενιαία κοινωνική πολιτική, αδιάρρηκτη. Λόγω του ότι απουσιάζει η κυρία Κόρχολα που είναι σκιώδη συζήτρια, μπορώ να την εκπροσωπήσω. Και ε, γι' αυτό λοιπόν ε, παρουσιάζω την, <clears throat> τον πίνακα ψηφοφορίων της δικής μας πολιτικής ομάδας. Ήθελα να πω ότι συνεργαστήκαμε με την κυρία Κόρχολα και με την κυρία Συγήτρια εδώ και πολλές εβδομάδες ε, με τρόπο αποτελεσματικό. Two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 μας ανακοινώσετε εάν και κατά πόσον αντικαθιστάτε κάποιον πρέπει λοιπόν να υπάρχει ενημέρωση για το ποιοι ψηφίζουν και ποιοι όχι. Δεν έχω πρόβλημα αν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν διαφωνούν στο να ψηφίζετε όλοι. Εγώ το ανακοινώνω, διότι θα έπρεπε κανονικά μας το κοινοποιήσετε. Παρακαλώ να πω ότι υπάρχουν περισσότεροι Πορτογάλες στην αίθουσα και να σας πω ότι εγώ εκπροσωπώ την πολυπληθέστερη πορτογαλική ομάδα. Το λέω προς τον συνάδελφο Κάστρο, διότι έχουμε στις πλήν των τυχερών παιγνίων. Κύριε Χάρμπορ, εσείς προτείνατε να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας προσπαθήσουμε. Εντάξει. Ξεκινάμε. Τροπολογία του κ. Μαρουμάτη, ψήφι πέρα. Περθμόν 4. 4 τροπολογία. Κοιτάξτε, οι πρώτες ε, έχουν εγκριθεί. Έπρεπε να το έχω καταστήσει σαφές. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές, σας. επαληθεύσουμε. Πέρα ψηφοφορίες. 28 υπέρ, 13 κατά. Παρακαλώ πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε την καταμέτρηση σωστά. Εντάξει, μπορεί να είστε κουρασμένοι, αλλά αν σηκώνετε τα χέρια θα πάμε γρήγορα. Ψήφινη ψηφοφορία 5 τροπολογία υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι τα 1, 2 και 3 εγκρίνονται. Πάμε στην τροπολογία 12. Α, απορρίφθηκαν, απορρίφθηκαν. Τροπολογία 12. Ψήφι πέρ. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έχει ψηφοφορία 26 υπέρ 15 κατά. Δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά. Δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ κατά. Επαλήθευση. Mm. 32 υπέρ 11 κατά. Προπολογία 16 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 18, 19 και 20. Όχι, καταπίπτουν. Περνάμε στην 21. ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 και 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μερικοί δεν ψηφίζουν και είναι δύσκολο. Για μας σε επαληθεύσουμε. 26 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Από εδώ πάντως ε, δεν είναι ξεκάθαρο, παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά εποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 3 υπέρ α, ε, χωριστή ψηφοφορία από το Highlight and Services έως το Consumer Design. Ψήφι υπέρ του πρότυματος κατά δεκτό, κατά συγγνώμη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Α, πάλι θέλουμε εντάξει. Yeah, it's 25 to 18, so it... 25 υπέρ 18 κατά. Δεκτό. 47. Ψήφι υπέρ. Α, και εδώ χωρίς την ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψήφι Κατά. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι κατά δεκτό. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 55 τροπολογία. Και εδώ χωρίς τη ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα ψηφιπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά έλεγχος έληξη ψηφοφορία 14 περί 27 κατά. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 68 υπέρ Στο κατάλογο παρατήρη πρόεδρος αναφέρεται το 5. Λοιπόν, εμπέσχετο θα ψηφίσουμε 68 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 και 70 ομού υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α, επαλήθευσης 24 ψήφοι κατά, 18 υπέρ, απορρίπτεται. Παράγραφος 5, 73 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74-78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ Εβδομήντα εννέα, διότι δεν θα κατέβησε Ψήφι υπέρ, κατά, επαλήθευση. Έλεξη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτό. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτή. Συμβαστική 8 προφορική τροπολογία προσθήκη του κ. Μάντερ. νομίζω ότι έχετε αντίγραφο Καλή την Επιτροπή κλπ. κλπ. ψηφι υπέρ τη προφορικής τροπολογίας προφορική τροπολογία Μάντερ. ψήφι κατά εγκρίνεται τροπολογία του Μπον προφορική και ευθεροπολογία ψήφι πέρ, κατά νομίζω πως εγκρίθηκε θα την επαληθεύσουμε όχι όχι γιατί οι, πολιτικές, οι μεγάλες πολιτικές μάδες υπερψήφισαν 85 υπέρ ε, συγγνώμη 8 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή 96 τροπολογία ψήφι κατά δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 τροπολογία Ψηφιπέρ, υπέρ κατά αποχές απορρίφεται, 108 110-111 ψηφιπέρ κατά αποχές 10 απορρίπτονται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108, 109, 111 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 112 Γκελάκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 του κ. Αγγελάκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή Εγκρίναμε την 112. Την 12, συγγνώμη. Συγγνώμη. Διάζομαι, αλλά βλέπω ότι τα καταφέρνονται. Προπολογία Μάντρες, υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. Παράγραφος 15. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτερη. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή Παράγραφος 18, 139, 140 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 15 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται, 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε καλού κακού. 26 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, δεκτή. 144 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 147 ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 148 το κύριο Γκέλακα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 149 ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός παρακαλώ That is mm. 32 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια, κυρία εισηγητρία. Yes. Did you want to say something now, Malcolm? Uh, well, just, I mean, I just repeat what... Όπως είπα και πριν, θα θέσουμε στη διάθεση όσων επιθυμούν την έκθεση της μειοψηφίας για να την υπογράψουν. Θα στείλω και ένα αντίγραφο στην κυρία Σάντε Μόζερ. Είναι σημαντικό το εγχείρημα που κάνει η Επιτροπή μας για την ανάπτυξη πολιτικής και στο εθνικό επίπεδο των κυβερνήσεων δηλαδή και στο ευρωπαϊκό. Εγώ επιθυμώ να συγχαρώ την Κρίσταλ για την καλή συνεργασία που είχαμε και βέβαια να διαβάσουμε πρώτα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δηλαδή όπως έχει προκύψει το κείμενο και μετά εξετάζουμε το κείμενο της μειοψηφία. Εγώ επιφυλάσσομαι πάντως σχετικά με την ψήφο μου στην Ολομέλεια. Θέλω πρώτα να δω το κείμενο όπως προκύπτει από την ψηφοφορία. Και ε, το ψήφισμα πάντως της μειοψηφίας θα πρέπει να απηχεί την σημερινή ψηφοφορία. Πρόεδρος, θα ε, σας διαβιβάσουμε το κείμενο όπως προέκυψε από την ψηφοφορία και μπορείτε να το εξετάσετε. Κύριος Μάντερς και εγώ συγχαιρώ την Κρίσταλ αλλά και την Επιτροπή ΙΜΚΟ διότι βλέπετε όταν εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη ένα επίμαχο θέμα ότι αναπτύσσονται διαφορετικές απόψεις και γνώμες και αυτό είναι ο λόγος που βρισκόμαστε και εδώ. Χαίρομαι λοιπόν που βάλαμε αυτό το επίμαχο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας. Κύριε Γκέπχαρτ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την Κρίσταλ για την εξαιρετική συνεργασία που μας προσέφερε και το τελικό αποτέλεσμα σε τόσο επίμαχο θέμα δείχνει πόσο ε, ισορροπημένη ήταν η εργασία της. Και γι' αυτό, το τονίζω αυτό άλλη μια φορά, και σε αντίθεση με αυτά που λέει ο Μάλκομ Χάρμπορ, είναι πολύ ισορροπημένη η εκθεσή της και νομίζω ότι την εξετέλεσε θαυμάσια. Mr. Ribeiro Castro, we're going to have a big debate now on gambling. Let's continue. Ευχαριστώ. Απλώς να πω ότι είναι ισορροπημένη η έκθεση και ελπίζω η μειοψηφία να προσεγγίσει την πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων και οικογενειών. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ σκόπιμο να γίνει αυτή η σύντομη ανταλλαγή απόψεων για να δούμε πώς θα κινηθούμε και στην Ολομέλεια. Λοιπόν, επόμενο θέμα, επόμενη ψηφοφορία. Ε, κύριε Μάντερς, νομίζω ότι είναι η δική σας έκθεση για την προστασία των καταναλωτών στην χρήση βιντεοπαιχνιδιών. Θέλετε κάτι να πείτε πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες που υποστήριξαν αυτή την έκθεση και νομίζω ότι φτάσαμε σε συμβασμούς παντού. Δεν χρειαζόμαστε επιπρόσθετη νομοθεσία, απλώς περισσότερες πληροφορίες και να προστατεύσουμε τους ανηλίκους πρωτίστως. Αυτό είναι ο απότερος στόχος και ελπίζω να τον επιτύχουμε με την έκθεση αυτή. Θα ήθελα το κοινό όσο αποχωρεί να μην συζητά μέσα στην αίθουσα αλλά εκτός αίθουσας. Λοιπόν, Επιτροπή Πολιτισμού 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Οι δύο επόμενες καλύπτονται. 1 της κυρίας Ματσούκα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2 απορρίπτεται. δύο Αγγελάκας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Της κυρίας Ματσούκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, έξι ε, 6 μάντερς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ Α, ναι, προχωρώ πολύ γρήγορα, με συγχωρείτε. 7 κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 τμήμα 1 ως προσθήκη υπέρ εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λίμπε δεν την ψηφίζουμε ούτε του πολιτισμού την 5 8 τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 τμήμα, α με συγχωρείτε, του κυρίου Αγγελάκα, την ξεχάσαμε 8, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 5 τμήμα 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, λίμπε 3 δεν ψηφίζεται, 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 9 του κυρίου Αγγελάκα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Λίμπε 13 και 5 δεν τις ψηφίζουμε, 12 τμήμα 1 ψηφίζουμε της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 είναι η επόμενη. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 ως προσθήκη της κυρίας Ματσούκα εγκρίνεται 2 τροπολογίες συμβιβασμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 Αγγελάκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, προήμιο α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 προήμιο 1 νομίζω ότι εγκρίνεται Α, τι κάναμε, το εγκρίναμε. Το α, το ένα συγγνώμη, υπέρ. Της Επίτροπης Πολιτισμού, το ένα, υπέρ. Μα δεν εγκρίναμε το τμήμα 1. Α, τότε καταπίπτει. Ωραία, δεν το ψηφίζουμε. Τελική ψηφοφορία. Ας γίνει ηλεκτρονικά. Για να δω τι παραμένει από τα θεμέλια. Πρέπει να ψηφίζουν 36. Πέρασε. Α, 35, 35 υπέρ, ομοφωνία και καμία εποχή. Πολύ ωραία κύριε Μάντερ, συγχαρητήρια. Yes. Yes. Darf ich nur damit es για να μην υπάρξει μετά καμία σύγχυση, θέλω να επισημάνω ότι κατά την φωτοτύπηση έγινε ένα λάθος. Στην σελίδα 10 λοιπόν παρακαλώ οι συνάδελφοί μου να κοιτούν τι κάνει η Κατρίν και εγώ. Θα δώσουμε λοιπόν τότε το σωστό σημάδι για την στάση που πρέπει να, ψηφι... να τηρήσουν στην ψηφοφορία. Κύριε Ανέρης, εσείς Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όσους συνεργάστηκαν γύρω από αυτό το θέμα, κυρία Φουρτού και άλλους, καθώς και τους βοηθούς και τη γραμματεία, διότι είναι γεγονός ότι αυτή η έκθεση, η πρόταση οδηγίας αλλάζει το κανονιστικό πλαίσιο, δεν ήταν απλή, αλλά λάβαμε υπόψη όλα τα στοιχεία και σκεπτικό έτσι ώστε να φτάσουμε σε έναν εύλογο συμβιβασμό. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τους πάντες διότι εξ αρχής ξέραμε ότι δεν ήταν απλό το θέμα αλλά αντιμετωπίσαμε όλες τις προκλήσεις. Okay, colleagues, if you'd like Σύντομες παρεμβάσεις παρακαλώ Μία φράση μόνο. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Νερίς και τους συνεργάτες της για την εργασία που ε, επετέλεσαν και που μας προσφέρει μια καλή βάση. Πρόεδρε, Μυστικώς υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τα πράγματα δεν είναι ιδεώδη βέβαια όπως τουλάχιστον είχα φανταστεί στην αρχή. Πάντως υπάρχουν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες εκφράζουν μια κοινή θέση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και ευχαριστώ όλους και όλες για τη συνεργασία τους. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ωραία. Άρθρο 1 λοιπόν. Θα το θέσω σε ψηφοφορία. Υπάρχει να των τροπολογιών, ψήφι υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2, ε, άρθρο 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. «109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έτσι δεν είναι, ναι. Και <clears throat> το 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 έχει αποσυρθεί, 89 έχει αποσυρθεί, ήτρε 5 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, νομίζω. Βέβαια, όλοι έχετε κουραστεί λίγο και δεν σηκώνετε καλά τα χέρια. Αν θέλετε επαλήθευση μπορούμε να κάνουμε δεύτερο τμήμα 12 υπέρ 26 κατά. κάτά, λοιπόν απερίφθη. Ήτρε 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 νέρις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ...95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 έχουμε ήδη συμφωνήσει έχουμε ήδη εγκρίνει την 87 και είναι ταυτόσιμες ας την ψηφίσουμε λέει η πρόεδρος καλύτερα 112 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχει αποσυρθεί 103 και 113 α πρέπει να την ψηφίσουμε ψήφι υπέρ ναι κατά αποχές εγκρίνεται 104 Handslick υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Χαντσλικ 105 υπέρ κατά αποχές όχι κατά κατά ακόμα Καλά, καλά. Ας επαληθεύσουμε 105. 13 υπέρ, 25 κατά. 106 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρα 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Θέλετε απολύθευση. 18 υπέρ 19 κατά. 108 και οι 38 μαζί υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Για το άρθρο 5. Αρκετές σελίδες βέβαια πιο κάτω. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Όλες οι υπόλοιπες εκπίπτουν. Συμβαστική 12 τώρα. Για το άρθρο 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Ακολουθεί η 25 για το άρθρο 7. για τη χρήση του σήματος ή Κατά. θέλετε επαλήθευση. Καλώς. υπέρ 21 κατά 17 εγκρίθηκε 168, 69, 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεν ψηφίστηκε 167 26 υπέρ κατά επαλήθευση υπέρ 21 κατά 17 εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ. Υπέρ ήτρε 17. Κατά. Απορρίπτεται. Λυπούμε και έτσι σε τι να κάνουμε. 174 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 176 υπέρ κατά όχι θα κάνουμε παρήθευση για το άρθρο 8 ε, 176 πέρας 18 υπέρ 20 κατά απερίφθη λοιπόν και αυτή Ήταν 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 Νιούτον ήταν υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά ας επαληθεύσουμε. Γιατί όπως είπα ορισμένοι δεν σηκώνουν καλά τα χέρια τους. «26 υπέρ 13 κατά». 181 εκπίπτει. «Ήτρε 19 υπέρ κατά». είναι ασυνήθιστη εικόνα που παρουσιάζει η ψηφοφορία. Ας επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται πάντω. Όχι, απερίφθη. 18 ε, υπέρ 20 κατά. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι υπόλοιπες. 190 υπέρ κατά ε, παρήθευση. Ίσως είναι καλύτερα, πιο γρήγορα δηλαδή. 19 υπέρ 20 κατά. Απερίφθη λοιπόν. Τροπολογία Χάντσλικ υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Δεκαεννέα υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται. Χάρμπορ 192. Ας ψηφίσουμε, ας επαληθεύσουμε η κατευθείαν δηλαδή ηλεκτρονικά. 18 υπέρ 20 κατά. 193, ας κάνουμε το ίδιο καλύτερα, ηλεκτρονικά. Δεκαεννέα υπέρ 20 κατά. 194. Ηλεκτρονικά λοιπόν. 18 υπέρ 19 κατά. Η τύχη με μία ψήφο διαφορά. Υποχρώσεις εισαγωγέων. 195. Άθρο 13 τώρα. 30. Νέρης υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Ας κάνουμε επαλήθευση. Υπέρ 21, 17 κατά. 198 υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί οι διαφορές είναι πολύ μικρές. 19 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Εναρμονισμένες προδιαγραφές. 199 κυρία Νέρης υπέρ και αυτό ηλεκτρονικά. 21 υπέρ 17 κατά. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207. Σβάπ. Υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Απορρίπτεται. Εγώ έχω βγάλει την ψήφο μου. Έχω αφαιρέσει την ψήφο μου. Λέει η πρόεδρος. Όπως είπα 18-21. 209. Α, ωραία, στην υπέρ. Ψήφι υπέρ, λοιπόν, εγκρίνεται. Άρθρο 17. 210 φουρτού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 18. 211 ρούλια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Υπέρ 22-16 κατά έγκρινεται. Άρθρο 19. 215 κάρας υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.18 Πλεσίνσκα υπέρ. Εγκρίθηκε. 218 λοιπόν υπέρ. Επαλήθευση καλύτερα ηλεκτρονικά. 19 υπέρ, 20 κατά. 217 υπέρ. Ας απολυτεύσουμε και αυτό ηλεκτρονικά. ...18 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται. 219 φουρτού υπέρ. Ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Α, 5 υπέρ και 34 κατά. Σαφέστατη διαφορά. 220 υπέρ. Κατά. Μόνο 5 ήταν υπέρ. Υπέρ λοιπόν τη 220. Α, μάλιστα έτσι καλύτερα. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Νερίς υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Άρθρο 20. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 224. Σφάμπ υπέρ. Επαλήθευση. 224. Πέρας. Α, 20 υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται. Ήτρε 22 δεύτερο τμήμα. Υπέρ, μάλλον ε, ηλεκτρονικά και αυτό. Ήτρε 22 δεύτερο τμήμα. 19 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται. Η 225 έχει αποσυρθεί. 22 τμήμα 3. Αλλά ας το κάνουμε ηλεκτρονικά. Α, είστε όλοι κατά. Καλά. Απορρίπτεται λοιπόν. 226 νερίς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 234 νταν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρθρο 22 235 πλεσίνσκα υπέρ Ω, δεν το ψηφίζουμε αυτό 23 236 υπέρ εδώ όμως θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπέρ 19 κατά 20. Ήσασταν κατά κύριε Μάντερς. Α, είστε υπέρ. Α, και πάλι τότε όμως ε, απορρίπτεται διότι είναι ισοψηφία. Τέτοιου δημοκρατία επιβάλλω εγώ εδώ από την έδρα του Πρόεδρου. Μάλιστα. 24-237. Ηλεκτρονικά. Ναι, ναι, ναι. 237. Επαλήθευση. Λειτουργεί το μηχάνημα τώρα κύριε Μάντες. 14 υπέρ 26 κατά απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 246 τώρα έτσι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 24 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε για να είμαστε πιο σίγουροι. Είκοσι υπέρ 19 κατά. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 37 υπέρ. υπέρ λοιπόν κατά επαλήθευση καλύτερα. «20 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται. 250 πλεσίνσκα υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 νέρις υπέρ, κατά. Ας, ας επαληθεύσουμε καλύτερα. 20 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. Είτε 25 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται νομίζω. 251 φουρτού υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.55 ρούλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά επαλήθευση α απορρίπτεται 256 υπέρ ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 20-19 εγκρίνεται. 2-57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 269 νέρις υπέρ. Επαλήθευση παρακαλώ. 21 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. 42 έχει αποσυρθεί. 2,71 ρούλε με ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα ωστόσο έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο. Ψήφι υπέρ. Επαλήθευση παρακαλώ. 26 υπέρ 13 κατά. 272 φορτού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 273 υπέρ. δεύση παρακαλώ. 273 handstick. 20 υπέρ 20 κατά ισοψηφία απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.75 μπρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.76 σφάπ υπέρ επαλήθευση παρακαλώ. Δεκατρεις υπέρ 26 κατά. Ήτρε 31 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 51. 277 Πλεσίνσκα υπέρ κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. ...17 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται... ...τροπολογία φορτού 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται... ...άρθρο 53, 279 νερίς υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται 2.80 υπέρ. Εγκρίνεται. 2.81 κάρας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράρτημα 1. 2.82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 283 κρέμερς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Ήτρε 32 εκπίπτει. 284 κρέμερς υπέρ κατά Επαλήθευση παρακαλώ. 2,84. Ισοψηφία 20 προς 20. Ήτρε 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,90 υπέρ Επαλήθευση παρακαλώ. Πρεστίνσκα Σουάμπ. Ισοψηφία 20 προς 20 απορρίπτεται. 2.91. Επαλήθευση. Είκοσι υπέρ 19 κατά εγκρίνεται. Ήτρε 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 45 ενεργείς υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά σε επαληθεύσουμε. Μάλιστα, 22 υπέρ 18 κατά. 46, ας την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. υπέρ 25-14 κατά. Τροπολογία Νιούτον ήταν 2,92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,93 Νιούτον ήταν υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται. 47 νερίς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 νερίς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 38 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρε 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 νερής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.97 έτσι δεν είναι. Και ή 42 που είναι ταυτόσιμες. Τις ψηφίζουμε όλες μαζί ψήφι υπέρ κατά. Επαλήθευση. Ναι επαλήθευση παρακαλώ. Καλό αργά παρά λέει η Πρόεδρος. 23 υπέρ 18 κατά. Ήτρε 1. Αιτιολογικές σκέψεις. Ήτρε 1 λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα νέρι, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε παρήθεση, Καλώς. Δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας. Υπέρ 19, 21 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 49 δέλτα πλεσίνσκα υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 50 νερίς. Θέλετε επαλήθευση. Καλώ. Επαλήθευση 49. Πλεστίνσκα. Απορρίπτεται λοιπόν. 24 κατάρα απορρίπτεται. Νέρις 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Αποσύρεται 51 κρέμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 χάρμπορ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 σβάμπ υπέρ Ας την ελέγξουμε 53 έλεγχος 21 υπέρ 20 κατά Άρα το ΕΛΚΑ έκανε τη διαφορά συσπηρώμενο έκανε τη διαφορά. 55. Χάνσλικ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 56. Χάρμπορ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57. Σβάμπ αποσύρεται. 58. Σβάμπ Ζίνσκα εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 17. Τρεις τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 60 αποσύρεται 61 Χάνσλικ υπέρ Α, αποσύρεται και αυτή. Δεχτήκαμε τις τρεις, άρα 62 Χάνσλικ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 Χάνσλικ υπέρ. Κατά Ας ελέγξουμε την 63. Ας ελέγξουμε την 63. 21 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται με μία ψήφο. 5 νέρις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 Χάνσλικ υπέρ. Θα την ε, ελέγξω. Την 64. Χάνσλικ, 64 ελέγχουμε. 22 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 8D και 67D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 23 στο 23, Νέρις Ρούλε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 69 Χάρμπορ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 Νέρις υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 70 Μπρι είναι προσθήκη υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 12 νέρις υπέρ, κατά. Μπορούμε να ελέγξουμε τη 12. Ελέγχουμε την 12 ηλεκτρονικά. 21 υπέρ και 20 κατά. Άρα εγκρίνεται κατά μία ψήφο. 71 νέρις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 αποσύρεται, 14 Νέρι υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, 73 Πλενσίνσκα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, 74 Πλενσίνσκα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, 75, 76 και η τρετρία υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνονται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά σα παρακαλώ. No, I am one of us. You can take me It's okay. 27 υπέρ 27 υπέρ κανένας κατά και 13 αποχέ. 14 απόχέ τελικά 28 υπέρ τελικά, 28 υπέρ. Θα είμαστε πολύ σύντομοι στην επόμενη ψηφοφορία. Έχουμε την απαλλαγή. Μπορούμε να έχουμε ψηφοφορία unblock. Πολύ καλή ιδέα. Θέλετε κάτι να πείτε? unblock. Γιατί δεν υπήρχε αμφισβήτηση υπέρ των έξι παραγράφων, υπέρ τελική ψήφος, υπέρ, άρα ομοφωνία και εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. πρόεδρε, για μία φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς για την εξαιρετική εργασία, λέει η βουλευτής. Γιατί είναι δύσκολο με τη δική σας ταχύτητα, ε, κυρία Πρόεδρε. Είναι άθλος. Νομίζω ότι οι διερμηνείς πάντοτε εργάζονται καλά, όχι μόνο όταν διερμηνεύουν εμένα.